Θα να ενημερώσω το σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 231 παραγραφός 4 του κανονισμού δεν ε, έχουμε λάβει κάποιο αίτημα για διευκρίνηση οπότε εγκρίνεται η σχετική διόρθωση. Το άρθρο 105 παράγραφος